αυτές οι τροποποίησεις της σύνθεσης των Επιτροπών. Από το Συμβούλιο έχω λάβει πέντε θέσεις του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την ε, ευνόηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών με την ε, απλοποίηση των δημοσίων εγγράφων. Δεύτερον, τον κανονισμό σε σχέση με την Ευρωπόλ. Τρίτον, την οδηγία σε σχέση με τις συνθήκες εισόδου και διαμονής των υπηκόν ε, υπηκών τρίτων χωρών. Τέταρτον, τον κανονισμό για, τα, για την προστασία των δεδομένων και την οδηγία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων. Οι τίτλοι αυτών των εγγράφων θα ανακοινωθούν στα πρακτικά αυτή τη Ολομέλειας. Το Κοινοβούλιο έχει στη διάθεσή του τρει μήνες για να εκφράσει γνώμη σε σχέση με την κοινή θέση του Συμβουλίου, ξεκινώντας από αύριο 12 Απριλίου 2016. Η Νομική Επιτροπή έχει λάβει θέση για δύο ε, κείμενα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο με διορθωτικά κείμενα. Βάσει του άρθρου 231, εάν μέσα σε 24 ώρες υπάρξει μια αίτηση από μια πολιτική ομάδα ή 40 μέλη του Κοινοβουλίου, θα τεθεί η γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής σε ψηφοφορία. Αλλιώς θα θεωρηθούν εγκεκριμένα.